Okay, friends, we start this meeting uh, a couple of minutes too late. Ε, συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε αργήσει λίγο. Ε, έχουμε πλήρες καθεστώς διερμηνία σήμερα, εκτός από δανέζικα, φινλανδικά, μαλτέζικα και κροατικά. Σημείο 2 ε, της σα διάταξη Ανακοινώσει της ε, Προέδρου. Ο πρώτο ε, τριμερής διάλογος για το Europass σε ό,τι αφορά τον κανόνα 55 θα λάβει λοιπόν χώρα στις 10 Οκτωβρίου από τις 7 έως τις 8.30 το απόγευμα. Με άλλα λόγια σήμερα λοιπόν το βράδυ. Και όπως Πολύ καλά γνωρίζετε. Ε, αργότερα σήμερα έχουμε μια κοινή δημόσια ακρόαση με την Επιτροπή ΚΑΛΤ σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οπότε θα χρειαστεί να μεταφερθούμε στην αίθουσα ESP 1G3 στις 3 ε, ε, σήμερα το απόγευμα. Αυτά λοιπόν και μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε όλοι σας τις κάρτες ψήφου σας. Μήπως θα πρέπει να περιμένουμε πέντε λεπτά ακόμα για να προσέλθουν όλοι και οι Οπότε αυτό θα κάνουμε. Πέντε λεπτά λοιπόν ακόμα. We'll Συνάδελφοι, θα περιμένουμε κανένα δύο λεπτά ακόμα. Γιατί βέβαια λόγω της ε, απεργίας ε, πολλοί συνάδελφοι χρειάστηκε να έρθουν με τα πόδια στο κοινοβούλιο. Οπότε θα σου δώσουμε πέντε λεπτά ακόμα. Συνάδελφοι, ελπίζω να έχετε βάλει τις κάρτες ε, μέσα στα μηχανήματα, προκειμένου να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία μας ε, ε, και ξεκινάμε με τη συμβαστική τοπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 20 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2. Συμβαστική τροπολογία 7. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 139. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ...151 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 152 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 153 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 155 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 156 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τοπολογία 7 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά σε ελέγξουμε ελέγχουμε την τροπολογία 7 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. Ας ξαναψηφίσουμε, συνάδελφοι. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν την ψηφοφορία μας για την τροπολογία 7. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με 22 ψήφους ε, κατά. Τη συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 167 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την τροπολογία 167 άρχεται η ψηφοφορία πέραση ψηφοφορίας απορρίπτεται με 24 ψήφους κατά. Τροπολογία 168 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 περ κατά αποχές εγκρίνεται 176 περ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά ας την ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 176 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας Απορρίπτεται με 25 ψήφους κατά. Συμβαστική τροπολογία 10 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 178 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 183 μαζί με την 184 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε και ηλεκτρονικά τις τοπολογίες 183 και 184. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας, απορρίπτονται με 25 ψήφους κατά. 186 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 187 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ας ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 11 ψήφι υπέρ ε, <coughs> συγγνώμη άρχεται η ψηφοφορία Πέρα τη ψηφοφορία απορρίπτεται με 24 ε, ψήφους κατά. 195 ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 196 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 200 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απο... εγκρίνεται. Τροπολογία 12 μαζί με την τροπολογία 215. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 204 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τοπολογία 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εκρίνεται. Τροπολογία 213 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 214 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 216 και 217 οι οποίε έχουν και δύο αποσυρθεί. Οπότε περνάμε στη συμβαστική τοπολογία 15 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 222 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 223 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά ας ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 231. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 μαζί με την τροπολογία 236. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε. Τις τροπολογίες 15 και 236 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. Περνάμε στην τροπολογία 239 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 18 ψήφι περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 240 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 242 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 251 υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται αλλά ας ελέγξουμε την 251 άρχεται η ψηφοφορία και πέρας και εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ περνάμε στην τροπολογία 252 ψήφοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 253 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά ας ελέγξουμε την 237 ε, άρχιτη ψηφοφορία πέραση ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά ας ελέγξουμε. Την 255. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Διαφορά 4 ψήφων. 256 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά ας ελέγξουμε την 263 άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε της ψηφοφορίας και πράγματι εγκρίνεται τελικά. 264 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 265 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 266 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 268 υπέρ, κατά αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε την 268. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας, όχι, δεν απορρίπτεται, εγκρίνεται με διαφορά μίας ψήφου. 269 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 270 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε την τροπολογία 272, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 274 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 274 άρχεται η ψηφοφορία και πέρας απορρίπτεται με 26 ψήφους κατά 276 ψήφι υπέρ ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται μάλλον αλλά ελέγχουμε την τροπολογία 276 άρχεται η ψηφοφορία πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 280 και 281 έχουν αποσυρθεί, οπότε περνάμε στην 285 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 286 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 289 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 290 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 291 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 19 ψήφι υπέρ Θέλετε να ελέγξουμε πρώτα την τροπολογία 293. Ηλεκτρονικά. Καλώς. Ελέγχουμε την 293, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με διαφορά δύο ψήφων. Συμβαστική τροπολογία 19. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 297 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 298 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 298 άρχεται η ψηφοφορία πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται διαφορά μιας ψήφου 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 1 ψήφι υπέρ ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 μαζί με την 35 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές Ας ελέγξουμε τις 2 ε, και 35, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. με διαφορά μιας ψήφου. Τροπολογία 36 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 36, γιατί δεν σηκώνετε καλά τα χέρια σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας και απορρίπτεται με διαφορά μια ψήφου. Η 37 καταπίπτει, περνάμε στη 38 ψήφι υπέρ. Α, όχι. Όχι, δεν καταπίπτει. Οπότε 37 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τροπολογίες 3 και 40. Ψήφι περ. ψήφι κατά, αποχές, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μια ψηφοδιαφορά. 39 καταπίπτει. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να γίνει έλεγχος σε τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 48 άρχεται πέρας Άλλη μια φορά ελεγχο ε, για τη 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 19 ψήφους. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται, τροπολογία 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται, 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται, τροπολογία 56, συγγνώμη, τι λέτε, να ελέγξουμε την 55. Άρχεται η ψηφοφορία για την 55. Πέρας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος της 56. Άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται 34 ψήφοι. Τρομάζω όταν καταλήγω σε, σε λάθη συμπεράσματα. 57 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 58 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 61 υπέρ κατά έλεγχος για την 61 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με 26 ψήφους 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την τροπολογία 63. Έλεγχος για την 63. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. Τροπολογία τώρα 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. έλεγχος για την 66 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτονται. τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 73 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τι είπατε? Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Εγκρίνεται. Ωραία, ξανά από την αρχή για την τροπολογία 73. Άρχεται η ψηφοφορία με την κάρτα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρεις ψήφοι διαφορά. Τροπολογία. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 78 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 79 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τοπολογία 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπ, Θα κάνουμε έλεγχο για την 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 106 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με τρεις ψήφους τροπολογία 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115 μαζί με την 116 διότι είναι ταυτόσιμες, υπέρ, κατά αποχές, εγώ θα έλεγα να γίνει ένας έλεγχος. Όσον αφορά την 115 και 116, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται με τρεις ψήφους διαφορά. Τροπολογία 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήταν σαφέστατο, θέλετε να διεξαχθεί έλεγχος για την 117. Τροπολογία 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 120 καταπίπτει, τροπολογία 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 123 υπέρ. Συγγνώμη, λέει πρόεδρος, τροπολογία 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 127 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 127. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 4 ψήφους. Τροπολογία 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 131 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Τοπολογία 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. Ευχαριστώ τον συγητή για το έργο που επετέλεσε. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε αμέσως. Σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Είναι το σχέδιο έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη-μέλη. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ρωμάνα Τόμς, την οποία όμως αντικαθιστά ο κύριος Κάσα. Θα δώσω μέσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Ντέιβιτ Κάζα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Um, Θα σας διαβάσω αυτό που μου έδωσε η κυρία Τόμς. Χτες μου το έστειλε. Ξέρετε ότι είναι ε, υποψήφια στις ε, προεδρικές εκλογές στη Σλοβενία. Τη ευχόμαστε καλή τύχη, παρόλο που θα προτιμούσαμε να μείνει εδώ, εν πάση περιπτώσει. Λέει ότι έλαβε 124 τροπολογίε στο σχέδιο έκθεση για την υλοποίηση πρωτοβουλία η κυρία Τόμψ ε, μας ευχαριστεί όλους για τις τροπολογίες μας αφενός και αφετέρου θέλει να ευχαριστήσει τους συμβούλους και τους άλλους συναδέλφους που βοήθησαν για να καταρτιστεί αυτή η έκθεση με την πραγματογνωμοσύνη τους. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες ενισχύουν πραγματικά το κείμενο, λέει η κυρία Τόμψ, οπότε πιστεύω ότι έχουμε καλή βάση για να εργαστούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και την ουσία, ε, να τονίσω και να σας εξηγήσω περί πρόκειται. Έχουμε υπογραμμίσει το πρόβλημα ε, να βρίσκουμε αξιόπιστες στατιστικές. Ε, η έκθεση βασίστηκε σε περιορισμένη πληροφόρηση. Δεύτερον, τονίζουμε ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν θα πρέπει να έρθει να αντικαταστήσει ούτε να υποκαταστήσει ε, τις εθνικές μεταρρυθμίσεις, αλλά είναι συμπληρωματικό εργαλείο προς αυτές. Εδώ έχουμε λάβει πολλές από τις τροπολογίες που προτείνουν ακριβώς το ίδιο. Τρίτον, τονίζουμε την ανάγκη να υπάρχει καλύτερο συντονισμός μεταξύ ε, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της αγοράς εργασίας για να υπάρχει μια αντιστοιχία της ε, ζήτησης προς την προσφορά και της προσφοράς προς τη ζήτηση. Επίσης, ε, θα πρέπει να εκπαιδεύονται καλύτερα οι άνεργοι, να φτάνουμε στους ανέργους με ειδικά μέτρα για την καταγραφή της ανεργίας και τον λεγόμενο needs που είναι οι ε, νέοι οι οποίοι είναι εκτός εκπαίδευσης, άσκησης, μαθητείας ε, και απασχόληση. Οι νέοι μας λοιπόν που αποκλείεται από την αγορά εργασίας θα πρέπει να έχουν ειδική αντιμετώπιση και ατομική πολλές φορές. Ε, στη συνέχεια, η ποιότητα της απασχόλησης είναι πολύ σημαντική. Αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα και οι νέοι θέλουν να έχουν ποιοτική εκπαίδευση, ποιοτική κατάρτιση και ποιοτική απασχόληση. Συχνά δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα όμως. Στη συνέχεια, τονίζουμε επίσης ότι απότερος στόχος της ε, πρωτοβουλίας ε, είναι η βιώσιμη θέση εργασίας. Θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία, επαναλαμβάνω. Το πρόβλημα είναι ότι τέτοια δεν διαθέτουμε και τα κράτη-μέλη δεν δίνουν τα στοιχεία και τα στατιστικά ε, σχετικά με τη βιωσιμότητα της απασχόλησης. Επίσης τονίζουμε την σημασία της βιωσιμότητας των κονδυλίων για την καταπολέμηση ε, της ανεργίας των νέων. Οι τροπολογίες που πηγαίνουν προς την κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουν την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ως βασικό ε, μηχανισμό χρηματοδότησης. Από τις τροπολογίες που λάβαμε υπάρχουν και πολύ καλές προτάσεις για το πώς θα βελτιωθεί η πρωτοβουλία αυτή στο μέλλον για την απασχόληση των νέων. Για παράδειγμα, να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε νέους που είναι σε ευάλωτες ε, ομάδες και καταστάσεις και να προσέξουμε περισσότερο τη διασυνοριακή αγορά εργασία. Σα ευχαριστώ και πάλι κυρία Τόμψ για τα σχόλια και τι τροπολογίε, σα ε, Λυπάτε που απουσιάζει και δεν θα μπορέσει να απαντήσει στι ερωτήσει, σα Ευχαριστώ. Η πρόεδρο, ευχαριστώ κύριε Κάζα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές, αρχίζοντας από τον κύριο Πενιφάη, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Κάζα που προσωπεί την εισηγήτρια την Κετόντς για την πολύ χρήσιμη αυτή εισαγωγή που έκανε και αυτά που ανέφερε. Συμφωνούμε εν γέννη, επιβεβαιώνεται ότι ακολουθήσαμε επικοδομητική προσέγγιση από την αρχή. Μαζί με συναδέλφους της ε, ομάδας μου ε, S&D υποβάλαμε διάφορες τροπολογίες ε, με στόχο ή να ενσωματωθεί να σωματωθούν στο κείμενο και να προταθούν κάποιες άλλες προτάσεις. Πολύ συχνά είναι αδύνατο οι τσιγητές να εξετάσουν όλα τα επιχειρήματα και να τα καλύψουν στο αρχικό κείμενο και λόγω περιορισμού, περιορισμένου χώρου και ανάγκες, ανάγκες μεταφραστικές. Ελπίζω η συνεισφορά της ομάδας μου και η δική μου να είναι χρήσιμες για να καλυφθούν κάποιες πτυχές όσον αφορά την αφορά στην αύξηση της προχρηματοδότησης Φερρυπίν, της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η πρόταση ε, της εκ των άνω συσσόρευσης πόρων ε, στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι κάτι χρήσιμο. Δράτω μας ευκαιρίες ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πάβελ που εκπροσώπησε τους σοσιαλιστές στην αποστολή που έγινε στη Σλοβενία και την Κροατία για την ενημέρωση που μας έκανε, που βοήθησε πάρα πολύ για την σύνταξη, την τελική των τροπολογιών. Είναι σημαντικό η Επιτροπή Απασχόλησης να καταληφθεί την ευκαιρία που μας παρέχει αυτή η έκθεση για να προωθήσουμε κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να, να επαναλάβουμε την υποστήριξη που παρέχουμε στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και την εγγύηση για τους νέους είναι βασικά εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ε, αν και δεν λύνουν τα προβλήματα, χρειάζονται περισσότεροι πόροι από τον υπολογισμό της Ένωσης και μετά το 2020 και μεγαλύτερες υποχρεώσεις που αναλάβουν τα κράτη-μέλη στο σύνολό τους για αυτό το θέμα. Πάνω θα είναι λιγότερο δαπανηρό να επενδύσουν σε αυτά τα εργαλεία σε σχέση με την απώλεια πλούτου που παράγεται από μεγαλύτερο αριθμό νέων που δεν εργάζονται. Θέλουμε να προτείνουμε κάποιες συστάσεις και συμβουλές για να χρησιμοποιούνται καλύτερα τα προγράμματα, παρουσιάζοντας μια φιλόδοξη συνεισφορά όσον αφορά τον ορισμό της ποιότητας των προσφορών. Είναι ένα θέμα πολύ βασικό ε, και πολύ αισθητό στα διάφορα κράτη-μέλη. Και τέλος θα πρέπει να καταγγείλουμε σαφώς την ανορθόδοξη χρήση των προγραμμάτων που πολύ συχνά χρηματοδοτήθηκαν μέσω της πρωτοβουλίας στην ενεργεία των καταπολέμησης της των νέων. Κάποια προγράμματα λανθασμένα, υπάρχουν καμιά φορά καθυστερήσεις στι πληρωμέ των νέων ή προσφορές με χαμηλή ποιότητα ή υπερβολική χρήση της περίοδου μαθητείας αντί πιο τακτική πρόσληψη. Όσον αφορά τι προσφορές, την προσφορά, έχουμε κάνει τροπολογίε για τα κριτήρια αξιολογήσεως που ξεπερνούν την απλή εξίσωση μεταξύ μέτρου που προσφέρεται και των αναγκών του υποψηφίου που πιστεύουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ περιορισμένος ορισμός. Ελπίζω ότι η συνεισφορά κατά των άλλων ομάδων ε, μέσω των προτάσεών τους θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε βιβαστικό κείμενο όσον αφορά αυτό το σημείο που ελπίζω να είναι φιλόδοξο και χρήσιμο για τους τελικούς χρήστες της εγγύσεως για τους νέους και για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Πιστεύω ότι το θέμα της ποιότητας είναι ένας κοινός στόχος να εγγυηθούμε ότι οι πολιτικές της Ενώσης στο πεδίο της απασχόλησης των νέων θα επιτρέψουν ταχεία και βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και να μην γίνεται εκμετάλλευση των πόρων λανθασμένη. Μετά θέλω να αναφέρω και μια άλλη πρόταση που υποβάλαμε να υπάρξει μια ε, γραμμή, αν θέλετε, hotline που ε, θα προτείνει τα διάφορα μέτρα για την ε, προώθηση, την επίλυση των προβλημάτων νέων. Ε, να μπορούν να το χρησιμοποιούν οι νέοι και άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι νέοι θα μπορούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Task Force, να καταγγέλουν λανθασμένη χρήση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ε, ταμεία, κυρίως όσον αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης καταγγελίας. Και η πρωτοβουλία αυτή για την απασχόληση των νέων εξάλλου είναι ένα άμεσο ε, μέσο που πρέπει να χρησιμοποιούν οι άνεργοι νέοι και δεν θα δίνει μόνο ποσοτική λύση όσον αφορά το πρόβλημα στα κράτη-μέλη και τα μέτρα που εφαρμόζονται. Ευχαριστώ λοιπόν για την πρόταση. Με τα χαρά να συνεργαστώ με τη συγκήτρια με όλε τι ομάδε, με το προσωπικό και του συναδέλφου για ε, τι επόμενε συζητήσει που θα γίνουν το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. και εγώ ευχαριστώ κύριε Μπενιφάη. Από την ομάδα η κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης, με χαρά παρακολούθησα το έργο της εισηγήτριας. Συμφωνούμε σε κάποια πράγματα για τη βελτίωση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Γι' αυτό οι δικές μας τροπολογίες υποστηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή και το πρόγραμμα ως εγγύηση για την νεολαία. Είναι δύσκολες οι συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη και η πρωτοβουλία αυτή ήρθε ως ε, αντίδραση σε μια επικίνδυνα υψηλή ενεργεία των νέων. Σε πολλές περιπτώσεις βοηθούν αυτά τα προγράμματα και ε, τα εργαλεία, αλλά δεν θα πρέπει να υποκρινόμαστε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και ελλείψει. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει προειδοποιήσει ε, ότι υπήρξαν πολλές απώλειες κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Θα πρέπει να λέμε και τα αρνητικά. Καλό είναι να αυξάνονται τα κονδύλια, να βλέπουμε και τι αξία έχουν τα προγράμματα. Δεν αρκεί η πολιτική βούληση και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό υποκατάστατο των εθνικών προσπαθειών και πρωτοβουλειών των κρατών μελών στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, την έρευνα, την καινοτομία. Αυτά είναι αρμοδιότητε των κρατών μελών. Υπάρχουν και μη κυβερνητικέ οργανώσει που θα πρέπει να συμμετέχουν καλύτερα στην εφαρμογή και στην υλοποίηση. Η εμπειρία μου λέγει ότι γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα η ΜΚΟ και πώς εργάζεσαι με νέους που είναι αποκομμένοι από την αγορά εργασίας. Καλό θα ήταν να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτές τις εμπειρίες. Τελευταία παρατήρηση είναι ανεπαρκή η προβολή και η διάδοση αυτών των πρωτοβουλειών. Οι νέοι, ιδιαίτερα αυτοί που αποκλείονται από την αγορά εργασία, δεν γνωρίζουν ε, τι δυνατότητε που του προσφέρονται ε, και ε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πάντως η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ καλή. Προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία με την εισηγήτρια και του σκιώδει εισηγητές και είμαι πεπισμένη ότι η έκθεση θα είναι τελικά μια επικοδομητική συνεισφορά. Ευχαριστώ. Thank you. I'll give the floor. Ευχαριστώ κυρία Λαμπάγεβα από την Ομάδα των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά τη Ρωμάνα Τόμτς για το σχέδιο εκθεσής της και τους άλλους σκιώδεις συγητές που έκαναν τις τροπολογίες. Πρέπει να πω ότι ήταν πολύ λίγες οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, διότι η εκθέση ήταν πολύ ισορροπή από την αρχή και τόνιζε τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά ή τα λιγότερο θετικά και τα προβληματικά σημεία της πρωτοβουλίας. Βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Οι δικές μου τροπολογίες ε, μιλούν για την ε, χρηστή διαχείριση των κονδυλίων αποτελεσματική αλλά και τα κίνητρα των νέων. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η πρωτοβουλία για έργα προσανατολισμένα στα αποτελέσματα και στη μακροχρόνια απόδοση. Όπως έχω πει επανελειμμένα, θα πρέπει να δούμε το, τη σχέση κόστος ωφέλειας και το μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Όπως είπε και η προλαλή σα, θα πρέπει να κοιτάμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, γιατί δεν έχει νόημα να συνεχίζεται χρηματοδότηση αν δεν υπάρχει αυτή. Επίσης, υποστηρίζω του συναδέλφου που ζητούν να συζητηθεί πρωτοβουλία αυτή στο επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο για να εξετάσουμε τη συνέχιση τη χρηματοδότηση του μέσου αυτού εφόσον μπορούμε πραγματικά να αποδείξουμε ότι πιάνουν τόπο τα χρήματα αυτά. Χαίρομαι για τη συνεργασία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε ε, στην ουσία των συζητήσεων και όλοι οι σκιώδεις ηγητές συμφωνούν ε, και είναι πολύ αγαστή η συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I can't see that, uh, madam. Ε, κυρία από την ΚΟΕ δεν παρευρίσκεται αυτή τη στιγμή αλλά είναι εδώ, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ. Ε, Τέρι, ε, ε, ε, χρειάστηκε να αγορεύσει στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, οπότε μου ζήτησε να σχολιάσω εγώ αυτή την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Η δική μας λοιπόν πολιτική ομάδα επέβαλε μία σειρά από τροπολογίες και εμείς εστιάζουμε κυρίως στο σοβαρό αντίκτυπο ε, ε, που έχει η ανεργία στην ε, φυσική αλλά και την πνευματική κατάσταση των νέων. Δηλαδή πραγματικά είναι καταστροφικές οι συνέπειες όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα κατά το οποίο παραμένει άνεργος ένας νέος τόσο πιο δύσκολο καθίσταται το να συγκεντρώσει περισσότερη εργασιακή εμπειρία στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν ο στόχο αυτή τη πρωτοβουλία είναι ακριβώ να φτάσει στου νέου, ειδικότερα του νέου εκείνου που είναι εκτό απασχόληση εκπαίδευση ή κατάρτιση, η καταρτιση οι επωνομαζομενη NEET, needs. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ακριβώ αυτού του ευάλωτου ε, νέου εκτό απασχόληση εκπαίδευση ή κατάρτιση, ε, ε, θα πρέπει να ζητήσουμε από τι αρμόδιε αρχέ απασχόληση των κρατών μελών να παράσχουν εξατομικευμένε υπηρεσίε σε αυτού του νέου και επίση να παρέχουν και εκπαιδευτικά ε, σεμινάρια έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη ε, ευαισθησία και από την πλευρά των ε, απασχολούμενων από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης σε αυτόν τον τομέα προκειμένου δηλαδή να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες αυτών των επαλωτών νέων. Αυτή η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα πρέπει να αποτελέσει την αρχή για μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα των νέων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκε του. Και η δουλειά αυτή που γίνεται σε ό,τι αφορά δηλαδή την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησή του, δεν θα πρέπει να σταματήσει σε καμία περίπτωση. Η μέχρι τώρα εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων έχει ε, καταδείξει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη εταιρική σχέσης προκειμένου να επιτύχει. Και γι' αυτό από τη δική μας πλευρά καταδικάζουμε το ε, ε, γεγονός ότι αυτή η, η εταιρική σχέση η οποία συμπεριλάμβανε τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους, τις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Ειδικότερα οι οργανώσεις δηλαδή της νεολαίας θα, πρέπει να, ε, έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό όσο και στην εκτέλεση και στην αξιολόγηση της ανλόγω πρωτοβουλίας. Ε, και τέλος, καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να ε, καταστήσουν πραγματικότητα τις ε, εγγύησεις για τους νέους. Θα πρέπει δηλαδή ε, να συνεχίσει το Κοινοβούλιο να λαμβάνει ενημέρωση και αναλύσει σε ό,τι αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Και επίσης καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν όλους τους ενδιαφερόμενους, όλους τους συναρμόδιους φορείς στην, στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτών των εγγύησεων για τους νέους. Ευχαριστούμε πολιτική από τους ε, Πράσινους και τώρα δίνω το λόγο στην Λάουρα Αόντια από το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για, αυτή την, ε, για αυτό το πρώτο κείμενο που μας υπέβαλε όσον αφορά την αξιολόγηση της χρήσης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Προτείνουμε αυτό το μέσο μια στιγμή που θεωρούμε ε, ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς εφαρμόστηκε στα διάφορα κράτη-μέλη η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ένα από αυτά τα μέσα είναι η εγγύηση για τους νέους. Λοιπόν, σε αυτή την πρώτη έκθεση θέλουμε να δείξουμε ότι η χρηματοπιστωτική οικονομική κρίση οδήγησε αύξηση της ανεργίας από 15% το 2008 στο 24% το 2013. Είναι ένα στοιχείο δηλαδή είχαμε σχεδόν διπλασιασμό αλλά θα πρέπει να δούμε ότι η ανεργία των νέων ποικίλει 10% το 2013 στη Γερμανία, Φερρυπίν στην Αυστρία και στην Ολλανδία ενώ σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Κροατία, η Ελλάδα εκεί έχουμε ποσοστά που πλησιάζει το 40%. Λοιπόν, το βασικό θέμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε οι εκθέσεις από τις διάφορες χώρες, από κάθε χώρα, για να μπορούμε να προβλέψουμε και διορθωτικά μέτρα για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας. Γιατί, διότι ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι οι διαφορές επιδόσεων οικονομικών και αναπτύξεως όσον αφορά την απασχόληση στις διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συμφωνούμε, Φερρυπίν, με τη σύσταση της συναδέλφου που προτείνει να επιταχυνθούν οι διαθωτικές μεταρρυθμίσεις για να μειωθούν οι διαφορές. Όχι διότι είμαστε κατά διαθωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά θα πρέπει να διερωτηθούμε ποιε μεταρρυθμίσεις διαθωτικές πρέπει να εφαρμοστούν. Αν η διαθωτική μεταρρύθμιση ε, ε ίσως δεν είναι καλή, ε, δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Στη, η ανεργία των νέων στην Ιταλία ε, είχαμε αρνητικά αποτελέσματα με λάθος μέτρα. Μια μετα, η μόνη μεταρρύθμιση που θα πρέπει να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη, κυρίως στην Ιταλία, είναι οικονομική, ε, αυξητική, επεκτατική μεταρρύθμιση που δημιουργεί ε, θέσεις επασχόλησης. Πηγαίνοντας στη Σικελία και στην Καλαβρία σε αποστολές, λίγο πολύ πριν από ένα χρόνο, για να δούμε πώς εφαρμόζεται η εγγύηση των νέων, είδαμε ότι η κατάσταση Δηλαδή ήταν δραματική, διότι δεν υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ στόχων που τίθενται από την πρωτοβουλία την απασχόληση των νέων με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Δεν υπάρχουν ε, ανοιχτά βήματα για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα μέτρο που μπορεί να γίνει διαθροτικό και αποτελεσματικό με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να μιλήσουμε για κατάρτιση, την κατάλληλη, τη σωστή. Δηλαδή να ληφθούν υπόψη ανάγκες των διαφόρων περιοχών και των επιχειρήσεων που μπορούν να απασχολήσουν νέους. Ε, αν δεν υπάρχουν, αν δεν ανοίξουν βήματα συζητήσεων, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών επιπέδων δεν θα τα πετύχουμε. Αυτοί που κάνουν την κατάρτιση δεν κάνουν τη σωστή ή αναγκαία κατάρτιση φερρυπίνη ή δεν την κάνουν καθόλου. Δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα να δίνουμε χρήματα στους νέους για την ε, κατάρτιση. Υπάρχει έλλειψη, κενό που είναι στη βάση κάθε πρωτοβουλίας που δρομολογείται και εφαρμόζεται. Ε, θέλουμε οικονομικές δραστηριότητες, κατάρτιση Θέλουμε ανάπτυξη οικονομική, κατάρτιση που έχει σαν στόχο την επίτευξη των σκοπών μας και να χρησιμοποιούνται σωστά τα διάφορα μέσα όπως είναι η πρωτοβουλία, η εγγύηση για τους νέους για να καλύψουν τα προβλήματα της ανεργίας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μην θεωρούμε ότι αν γίνει θετικό το μέτρο έχουμε βρει την αποκλειστική λύση για να λειτουργήσει για την εγγύηση των νέων. Η πρωτοβουλία για την αποσχόληση των νέων χρειάζεται συγκεκριμένα προγράμματα, σαφείς ιδέες, κυρίως συνεχής συζήτηση, παρακολούθηση και προσοχή. Οι πόροι μπορεί να υπάρχουν και ας είναι ανεπαρκείς. Αλλά όταν σπαταλιούνται ή χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, διαφορετικούς από αυτού που καθορίζονται στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, τότε έχουμε πλήρη χρεοκοπία των μέτρων. Άρα επιφυλασσόμεθα για τη συνεργασία μας με συνάδελφο Τόμκιν και τους διάφορους ε, συναδέλφους για να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το τελικό κείμενο. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Μαρτάν που προσωπείτε την ομάδα ΙΕΝΕΦ, παρακαλώ. Ε, όχι, ζητώ συγγνώμη για ε, την απουσία του δόκτωρο Μαλά που έχει μπλοκαριστεί στη Γαλλία λόγω των γαλλικών πια απεργιών, όχι των εδώ. Sí. Ευχαριστώ. You don't want to... Α, δεν θα πάρετε εσείς το λόγο εξ ονόματος της ομάδας σας για να αντικαταστήσετε τη δόκτωρα Μαλά. Ο κύριος Λαβριέ έχει ζητήσει το λόγο. Α, άλλος, ο κύριος Πάβελ. Ε, ε, ευχαριστώ. Σύντομα να σας πω δύο λόγια για το θέμα. Ε, εκτιμώ τη δουλειά των συναδέλφων πραγματικά και ιδιαίτερα στην αποστολή που είχαμε πάει στη Σλοβενία και την Κροατία ε, μπορέσαμε να δούμε ότι είναι αντίστοιχα τα προβλήματα που έχουν οι χώρες αυτές με τις δικές μας. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, πιστεύω, και μπορεί να γίνει με το συγκεκριμένο θέμα και την έκθεση, να βελτιωθεί το πρόγραμμα που έγινε όταν αποφασίστηκε για να απαντήσει σε μια έκτακτη ανάγκη. Αλλά να το συνεχίσουμε, να βελτιώσουμε την απασχόληση των νέων και πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ενημερώνονται εκείνοι που δεν ε, ψάχνουν πληροφορίες. Δεν είναι αρκετό να έχουμε σε μια ιστοσελίδα πληροφορίες για κάποια προγράμματα ή στις εφημερίδες. Οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι, δεν τις ψάχνουν, δεν τις διαβάζουν. Αυτούς πρέπει εμείς να τους βρούμε και να τους ενημερώσουμε και να πάμε την πληροφορία σε αυτούς, γιατί δεν πρόκειται να την αναζητήσουν οι ίδιοι. Αυτό είναι το θέμα με τα συγκεκριμένα προγράμματα. Πρέπει να συνεχιστεί το ίδιο πρόγραμμα, ίσως να αυξηθεί η πρικοδότησή του όχι βέβαια να υποκαθιστά ή να αντικαθιστά τα εθνικά προγράμματα, αλλά ε, να τα υποβοηθά, το χρειάζεται. Πολύ καλό το πρόγραμμα είναι, πιστεύω, και περιμένω να δω το τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος της αγορεύει βούλετε. Ο κ. Κάσα. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους παρόντες, Έλαβα υπόψη όλες τις συστάσεις και τα σχόλια. Θα διαβιβάσω στην κυρία Ρωμάνα Τόμιτς τα σχόλια. Δεν υπάρχουν επίμαχα ζητήματα. Άρα πιστεύω θα είναι πολύ καλή έκθεση και ευχαριστώ πολύ για τις συνεισφορές σας. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι κάποιοι εκπροσωπούν τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Η κυρία Κόλεβα ίσως η κυρία Κολέβα έχει το λόγο. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Να πω ότι αυτή η έκθεση πράγματι έρχεται την κατάλληλη στιγμή, είναι πολύ χρήσιμη. Διότι προετοιμάζουμε νέες προτάσεις για το πώς τα, ευρωπαϊκά διαθωτικά και επενδυτικά ταμεία θα υποστηρίξουν την απασχόληση των νέων. Δημιουργήθηκε αυτή η πρωτοβουλία για τους νέους ή την απασχόληση των νέων σαν ένα εργαλείο για τη χείριση κρίσεων. Αλλά τώρα επεξεργαζόμεθα πιο βιώσιμη υποστήριξη της πολιτικής για τους νέους μετά το 2020. Και έτσι σημειώνουμε όλες τις χρήσιμες συστάσεις της εκθέσεως. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα έχουμε ευκαιρίες να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ήδη αναφέρθηκε αυτό. Βέβαια, αυτή η ευρεία πρωτοβουλία δεν υπήρξε επιτυχή σε κάθε κοινότητα όλων των κρατών μελών. Όμως, υπάρχουν πολλά καλά αποτελέσματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. όταν ανακαλύπτουμε νέες μορφές για την εκπαίδευση των νέων ή για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αυτές θα είναι χρήσιμες. Που θα απορρέουν από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, όπως πολλοί αναφέρατε. Τα προβλήματα ήταν σοβαρότατα. Κάτι έπρεπε να γίνει. και προσπαθούμε να βρούμε καλύτερες λύσεις. Τώρα που η κατάσταση δεν είναι πλέον εκρηκτική στην αγορά εργασίας για τους νέους. Τουλάχιστον συγκρίση με το όταν ξεκινήσαμε. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου. Τούτου λεχθέντος έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα από το πρόγραμμά μας. Αλλά αν εκείνοι που χρειαζόμαστε είναι ήδη παρόντες, ας προχωρήσουμε. Πάμε στο σημείο 5 της σημερινής διατάξεως. Οικονομικά ωφέλη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. We are still waiting for... Περιμένουμε κάποιους mm. από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Η κυρία Λάμπακ δεν είναι εδώ. Oh. Είναι καθοδόν. Ευχαριστώ. Θα περιμένουμε πέντε λεπτά. Και μετά θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για τα οικονομικά ωφέλη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πεντάλεπτο διάλειμμα λοιπόν. Uh, yes, well, uh, we proceed with... Καλώς ε, συνεχίζουμε με το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή τα οικονομικά ωφέλη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ξεκινήσουμε δίνοντας ε, το λόγο στην κυρία Λάγκμπακ που είναι η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Θα μας κάνετε λοιπόν μία παρουσίαση ως προς πώς έχουν τα πράγματα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και με χαρά μου βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας κάνω μία παρουσίαση εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης. Δηλαδή ε, την ε, επιτροπή που βρίσκεται εγκύτερα ακριβώ σε αυτόν τον τομέα τη οικονομική και επαγγελματική ανεξαρτησία και στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του καθενό. Προτού όμω περάσω στην παρουσίασή μου, θα ήθελα να σα αναφέρω, ε, αναφέρω ποιες είναι οι κύριε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στον τομέα τη ισότητα ε, των φύλων και πώ επηρεάζει του άντρε και τι γυναίκε ε, τη σήμερα ημέρα και με διαφορετικό τρόπο. Αν δούμε για παράδειγμα το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά τα χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και την αποσύνδεση από την αγορά εργασία, ε, εδώ σας δείχνουμε λίγο και το τι έχουμε συγκεντρώσει ως στοιχεία, δηλαδή από διάφορους τομείς και με βάση διαφορετικές μελέτες και θα διαπιστώσετε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ότι ε, στους τομείς εκείνους όπου έχουμε χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης, οι γυναίκε, με χαμηλά δηλαδή ε, εκπαιδευτικά προσόντα, έχουν ε, πολύ μεγάλο κίνδυνο να αποκλειστούν από την αγορά εργασία και για μεγάλο ε, χρονικό διάστημα να μην ε, συμμετέχουν στο ε, εργατικό δυναμικό. Και διαπιστώσαμε σε μία μελέτη που κάλυψε 6 εκατομμύρια άτομα, 17% ε, των ε, ε, γυναικών που έχουν χαμηλά προσόντα δεν έχουν εργαστεί ποτέ και 2 εκατομμύρια άντρες ταυτόχρονα από την ίδια μελέτη και εκείνοι με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα δεν έχουν εργαστεί ποτέ τώρα. Εάν περάσω στις επόμενες προκλήσεις να σας πω ότι εξετάσαμε και ε, τις ε, μητέρες οι οποίες εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας. Εξετάσαμε δηλαδή εδώ το διαφορετικά, ε, τις συνθέσεις των οικογενειών. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχουμε πάντοτε ε, της, ε, την παραδοσιακή σύνθεση της οικογένειας, ειδικότερα ακριβώς επειδή υπάρχουν και περιπτώσεις οικογενειακής βίας και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες σήμερα ημέρα και το 85% αυτών είναι ε, μόνες μητέρες με παιδιά. Και αν δείτε εδώ την, την τελευταία στήλη βλέπουμε τη μεγαλύτερη διαφορά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Εάν έχουμε μια οικογένεια με τρία ή περισσότερα τέκνα, αυτή η σύνθεση έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά δηλαδή το κίνδυνο να μην εργάζονται οι γυναίκες αυτών των οικογενειών, ε, γονείς δηλαδή. Η διαφορά δηλαδή μεγαλώνει όλο ένα ε, και περισσότερο με κάθε επιπρόσθετο τέκνο. Δηλαδή το 55% βλέπουμε εδώ ε, μόνο των γυναικών οι οποίες είναι γονείς σε μια οικογένεια με τρία υπεραιτέρω ή περισσότερα ε, παιδιά. Αλλά κάναμε και μια περαιτέρω ανάλυση και αν ε, δούμε ε, τον κίνδυνο φτώχεια αυτών των γυναικών, από αυτό το 55% που δεν εργάζονται, το 44% κινδυνεύει να βρίσκεται κάτω από το όριο της ένδυας εάν ο άλλος γονέας της οικογένειας χάσει τη θέση εργασίας τους. Οπότε, εάν ή μάλλον κατά τη ε, διάρκεια της ε, χάραξης των πολιτικών μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό το πολύ σημαντικό ε, στοιχείο. Τώρα, έχουμε λοιπόν αυτούς τους μόνους αγωνίες και βλέπουμε στις διάφο στα διάφορα κράτη-μέλη πόσο διαφορετικές είναι και οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά δηλαδή και τις διάφορες ε, πολιτικές ένταξεις στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Πώς δηλαδή επηρεάζονται από αυτές τις πολιτικές μόνοι γονείς και είδαμε και στις υπόλοιπες μελέτες πόσο σημαντικό είναι να παρέχεται κοινωνική προστασία, ε, ειδικότερα ε, σε ό,τι αφορά ε, γονείς με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευση, γιατί εκεί ε, αυτοί οι γονεί έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν κάτω από το όριο τη φτώχεια. Επίση, βλέπουμε πω οι νέε γυναίκε και οι νέε με ε, παιδιά μικρή ηλικία είναι εκείνε ε, που εργάζονται λιγότερο από όλε τι υπόλοιπε κατηγορίε του εργατικού δυναμικού. Επίση, το 26% των μόνων γονέων και κυρίω των μόνων γυναικών γονέων έχουν χαμηλή ένταση εργασία. Δηλαδή, εάν συμβεί οτιδήποτε, Ε, δηλαδή μια νεαρή για παράδειγμα γυναίκα με νέα ε, παιδιά, όχι μόνο χάνει ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, αλλά αυτόματα και άμεσα περιέρχεται σε κίνδυνο να βρεθεί κάτω από το όριο της στόχιας. Μία ακόμα διαφάνεια τώρα σας δείχνω. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στον εργασιακό και τον ιδιωτικό βίο. Βλέπετε ένα από τα πορίσματα από τον ε, δείκτη για την ισότητα των φύλων, τον οποίο, για τον οποίο θα κάνουμε και μια δημοσίευση αύριο και διαπιστώνουμε εδώ πώς το φύλλο συνδέεται και με άλλα ε, χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, ο τύπος της οικογένειας, ε, το τρονικό υπόβαθρο και το καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ έναν πληθυσμό εδώ ατόμων ε, τα οποία φροντίζουν για παράδειγμα κάποια μέλη της οικογένειας μεγαλύτερης ηλικίας τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα. Τη βλέπουμε στην πρώτη εδώ κατηγορία, ε, ε, την οικογένεια δηλαδή εδώ, βλέπουμε πως το μεγαλύτερη, τη μεγαλύτερη διαφορά υπάρχει σε αυτούς τους μόνους γονείς. βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά δηλαδή σε ό,τι αφορά την εργασία που αφιερώνουν ε, σε ε, αυτές τις δραστηριότητε οι μόνοι γονείς, μόνοι άντρες και μόνοι γυναίκες και μετά βλέπετε και την ε, διαφορά που υπάρχει σε ό,τι αφορά την απόκληση, σε ό,τι αφορά τα, την χώρα γέννησης. για παράδειγμα τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα θα πρέπει να προβλέπετε σε ό,τι αφορά τη φροντίδα παιδιών ή άλλων ε, συγγενών. Οπότε βλέπετε με αυτόματα πόσο μειώνονται ε, τα, ε, οι δυνατότητες για την επιτυχία εξέβρασης της εργασίας. Επίσης, εξετάσαμε τις ε, πολιτικές απασχόλησης σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ ε, των φύλων και σε ό,τι αφορά τον τύπο παραγωγής. Και αν εξετάσουμε ε, τον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της πρόνοιας που θεωρούνται πως είναι, κυριαρχούνται κυρίως από τις γυναίκες και μετά τους τον άλλο τομέα των φυσικών επιστημών, θα δούμε ότι έχουμε δύο τελείως αντίθετους πόλους μεταξύ τους. Καθώς ο τελευταίος κυριαρχείται από άντρε. Για παράδειγμα, ε, ο, πρώτο, ο, πρώτος τομέας που ανέφερα, δηλαδή που κυριαρχείται από τι γυναίκε, υγεία, πρόνοια και ούτω καθεξής, έχει χαμηλότερα επίπεδα ε, μισθών. Ε, το 80% σε αυτό το τομέα είναι γυναίκες εργαζόμενοι. Και αν δούμε τις σχετικές μελέτες θα διαπιστώσουμε ότι οι άντρες λαμβάνουν υψηλότερου μισθού ε, από ό,τι ο μέσο όρο. Δηλαδή υπάρχουν άντρε οι οποίοι απασχολούνται σε αυτό το τομέα, αλλά ο αριθμό του είναι μειούμενο, δηλαδή των άντρων οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα. Αν δούμε από εκεί και μετά ε, ε, τον ε, αριθμό ε, των γυναικών οι οποίες ε, απασχολούνται στον τομέα των φυσικών επιστημών και γενικότερα στον τομέα STEM, στα τελευταία δέκα χρόνια το ποσοστό των γυναικών έχει παραμείνει σταθερό. Δηλαδή δεν παρέχονται περαιτέρω κίνητρα για την απασχόληση των γυναικών σε αυτόν τον τομέα STEM. Επίσης, αν δείτε εδώ την, τις κατηγορίες θα διαπιστώσετε ότι ο αριθμός των ανδρών στον τομέα της υγείας Εκπαίδευση και Ε, βαίνει μειούμενος γιατί ε, ε, το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των ανδρών που εργάζονται στο σχετικό ε, τομέα βρίσκεται στην ηλικία ομάδα των 60 με 64 που σημαίνει στο εγγύς μέλλον εντάξει, ίσω να μην πούμε ότι δεν θα έχουμε κανέναν άντρα που θα εργάζεται σε αυτό το τομέα, αλλά πολύ λιγότερου. τώρα, αν δούμε στου ε, επιμέρους τομείς εκπαίδευσης θα ε, διαπιστώσουμε πόσο μεγάλη είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα ε, σε αυτούς τους τομείς απασχόλησης. Για παράδειγμα, αν δούμε την εκπαίδευση, θα διαπιστώσουμε ότι μόνο το 18% των ανδρών σπουδάζουν ένα επάγγελμα εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Ε, και κυρίω ε, οι άντρε ενδιαφέρονται για το πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό τομέα και όχι τόσο πολύ για τα σχολεία. Και βέβαια και το στερεότυπο τη κοινωνία ε, του αποθαρρύνει από το να επιλέξουν ένα τέτοιο επάγγελμα. Αντιθέτω, στι φυσικέ επιστήμε βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τι γυναίκε για να σπουδάσουν αυτόν τον τομέα, αλλά εάν επιλέξουν τον τομέα των φυσικών επιστημών επιλέγουν ε, επαγγέλματα διδασκαλία, δηλαδή δεν ε, καταλήγουν τελικά σε ένα επάγγελμα ε, υψηλής, υψηλών απολαβών, για παράδειγμα έρευνα και ούτω Σε ό,τι αφορά τώρα τις τεχνολογίες ICT, έχουμε ένα, το ποσοστό 21% για τις γυναίκες οι οποίες σπουδάζουν σε αυτό το τομέα και γνωρίζετε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας. Με βάση δηλαδή τις προβλέψεις που έχουμε, ο εν λόγω τομέας είναι ε, εκείνος για τον οποίο χρειάζονται όλοι να έχουν επαγγελματικά προσόντα. Και μόνο λοιπόν το 1 πέμπτο του συνόλου των φοιτητών είναι γυναίκες, των φοιτητών δηλαδή οι οποίοι σπουδάζουν ακριβώς ε, ε το ICT. Και κάτι αντίστοιχο ισχύει και από το τομέα της μηχανολογίας, μεταποίησης και κατασκευής. Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τη συμφορή σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτά τα επαγγελματικά προσωπικά και πώς θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσει στο μέλλον. Κάτι συνέβη με την παρουσίαση. Άρα λοιπόν, ε, ότι οι σημερινέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιε και ε, διαπιστώνοντα ότι δεν ενθαρρύνουμε τι ε, γυναίκε να σπουδάσουν επαγγέλματα STEM και δεν ενθαρρύνουμε του άντρε να σπουδάσουν επαγγέλματα τομέα ε, υγεία, εκπαίδευση ε, και πρόνοια, ε, τα πράγματα θα δυσκολεύσουν γιατί πραγματικά αν το κάνουμε, αν ενθαρρύνουμε ε, την ενασχόληση ε, των δύο διαφορετικών φύλων με τους εκάστοτε τομείς θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα και σχετική μελέτη που κάναμε χρησιμοποίησαμε το μοντέλο E3ME e, το οποίο έχει σχεδιαστεί από το Πανεπιστήμιο του Κέμπτη σε την οικονομετρία και προσπαθήσαμε εδώ να εξετάσουμε από κοινού όλους τους ε, ε, τομείς πολιτικής και βλέπω πως έχει επιστρέψει εδώ ε, διαφάνεια στην οθόνη. Άρα λοιπόν αναλύσαμε όλα τα διαφορετικά σενάρια, όλους τους διαφορετικούς ε, τομείς και προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε εάν ε, γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα σε ό,τι αφορά δηλαδή τα επαγγέλματα ε, που κυριαρχούνται από γυναίκες ε, και υπάρχει εξίσωση σε αυτά τα επαγγέλματα όπω και τα επαγγέλματα που κυριαρχούνται από άντρες διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλοί απτά οικονομικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι αν υπάρξει επένδυση σε αυτή την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, αν αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα, αν επενδύσουμε στην ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου, αν δηλαδή αντιμετωπίσουμε με όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπήρχε σημαντικό οικονομικό όφελος, συγκεκριμένο οικονομικό όφελος και και εδώ σας δείχνω ποια είναι η βάση του υπολογισμού. Δηλαδή, ποιε είναι οι εξελίξει που λαμβάνουν χώρα σήμερα, λαμβάνοντα υπόψη και το ότι, ότι Ε, δεν θα ε, συνεπάγεται μια επιδίνωση της κατάστασης των ανδρών, αλλά εξίσωση των γυναικών με τους άντρες στους τομείς ε, όπου δεν έχουμε την επαρκή προσώπηση από τις γυναίκες. Άρα λοιπόν εδώ εξετάσαμε διαφορετικά σενάρια και τα στοιχεία στα οποία βασιστήκαμε αφορούσαν το σενάριο όπου εξετάζουμε καταρχήν ε, την ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ε, χάσμα μεταξύ των διαφορετικών φύλων. Να διαφυρώσουμε αυτό το χάσμα στην τριτογενή εκπαίδευση. Ήταν ένα από τα σενάρια και το άλλο ήταν η μη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό σε ό,τι αφορά δηλαδή τις μισολογικές διαφορές και ούτω καθεξής. Από εκεί και μετά εξετάσαμε την ίδια, τη, τις ίδιες τις μισολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων και επίσης καθώς μιλάμε συνέχεια για τη ε, γύρανση του πληθυσμού μας εξετάσαμε και τη δημογραμμική μεταβολή και το πώς δηλαδή μπορούμε να αυξήσουμε ε, και ε, τα σχετικά ποσοστά. Ε, τα ποσοστά λοιπόν λογονομότητας και προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τα ωφέλη λοιπόν αυτών των παραγόντων από κοινού. και βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια το αποτέλεσμα αυτού του πολύ σαφούς και αντικειμενικού υπολογισμού με βάση το οικονομικό ε, μοντέλο έως το 2050. Εάν λοιπόν γεφυρώσουμε αυτά τα χάσματα, εάν επενδύσουμε με ενεργό τρόπο στα σχετικά μέτρα, θα διαπιστώσουμε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κεφαλήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθεί κατά 9,6% χωρίς καμία περαιτέρω εκπαίδευση. Απλώς δηλαδή μέσω γεφυρώματος αυτού του χάσματος μεταξύ των φύλων. Ε, και σε, σε αριθμούς συγκεκριμένους το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται σε 3,15 εκατομμύρια ευρώ. Άρα εξετάσαμε από εκεί και μετά ε, ε, τα επιμέρου σενάρια ξεχωριστά. Είδαμε για παράδειγμα το τι θα μπορούσε να γίνει να κλείσει το χάσμα σε ό,τι αφορά το τομέα ε, STEM. Όπω είπαμε, ένα τεράστιο τομέα ε, όπου υπάρχει μια τεράστια ζήτηση για επαγγελματικά προσόντα. Εάν λοιπόν οι άντρε συνεχίσουν να σπουδάζουν στα ποσοστά που προβλέπονται κανονικά, χωρίς να υπάρξει μεταβολή, αλλά διασφαλίσουμε ταυτόχρονα ένα ενδιαφέρον από την πλευρά των γυναικών για σπουδές σε αυτό το τομέα, βλαπιστώνουμε ότι θα δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και αν αυτές οι θέσεις εργασίας καταλαμβάνονται κατά το 70% των γυναικών, θα φτάναμε στο αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ και έχουμε προβλέψει δηλαδή ένα γρήγορο σενάριο γρήγορης μετάβασης και ένα σενάριο ε, βραδύτερης ε, μετάβασης. Ε, σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ένα τεράστιο όφελος στο αργό αν θέλετε βραδύ σενάριο προσπαθούσαμε να διαπιστώσουμε τι θα συμβεί σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν προβούν σε πολύ σε επενδύσεις. Δηλαδή ε, σε περίπτωση όπου τα κράτη-μέλη αναλάβουν κάποια δράση συμπληρωματική προς αυτή που λαμβάνουν σήμερα. Και βλέπετε ποια είναι η διαφορά, ανάλογα δηλαδή με τα ενεργοποίηση των κρατών μελών. Εδώ βλέπετε μια διαφάνεια που αφορά συγκεκριμένα στο τέταρτο ε, σενάριο. Εάν δηλαδή ε, βελτιώσουμε την ισορροπία εργασιακού και ιδιωτικού βίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν κλείσουμε, γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ των δύο φίλων μόνο ε, με βάση τα, αυτά τα μέτρα θα γεφυρώνουμε αυτόματα και το, το, τη μισολογική διαφορά. Και βλέπετε εδώ και τι θα συνέβαινε σε επίπεδο ε, ποσοστών γονιμότητας, γιατί οι γυναίκες θα είχαν πλέον την αίσθηση ότι λαμβάνουν υποστήριξη, δεν θα αντιμετώπιζαν την κατάσταση που σας έδειξα προηγουμένως στη διαφάνεια των μονογονοϊκών οικογενειών με μία ε, γυναίκα ως ε, γονέα η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο να ε, βρεθεί κατά από το όριο τη Βλέπετε λοιπόν πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα σύγκριση με σήμερα. Ε, η βελτίωση δηλαδή σε ό,τι αφορά τα ποσοστά γονιμότητα. Ε, και από εκεί και μετά ε, έχουμε εξετάσει με βάση τον δίκτυο που όπως είπα θα παρουσιαστεί αύριο ε, το τι θα συνέβαινε στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε προβλέψει εδώ δύο διαφορετικά σενάρια με βάση δύο διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Και η ομαδοποίηση εδώ των κρατών μελών έγινε Ε, με βάση ε, ε, κατηγορία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της, του θεματολογίου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη ανισότητα των φύλων. Είχαμε δηλαδή 7 κράτη-μέλη με τι καλύτερε επιδόσεις, μετά μέτρες επιδόσεις και χαμηλέ επιδόσει. βλέπουμε λοιπόν εδώ το, την πλέον ομάδα η οποία είναι, έχει καλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων και βέβαια δεν θα χρειαστεί να επενδύσουν σε τόσο σημαντικό βαθμό, ακριβώς γιατί ήδη βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η ομάδα 1 θα μπορούσε να υποφεληθεί ε, τα μάλλα. Δηλαδή, αν έκανε τα όσα κάνει η ομάδα 3, θα μπορούσε να εξασφαλίσει έως το 2050 ποσοστά αύξηση του ακαθάριστου των χώρων όντως στη του 12%. όπως σας είπα έχουμε εξετάσει επιμέρους εδώ ε, ζητήματα και εξηγούμε βέβαια, ε, όπως αναφέρθηκε και στον ιστότοπό μας, ε, ακριβώς λεπτομερώς το μοντέλο και ανάλυση που έχουμε χρησιμοποιήσει. Ελπίζω λοιπόν να βρείτε τον χρόνο και τον ενδιαφέρον για να διαβάσετε αυτή τη μελέτη. Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας διαθέσουμε περαιτέρω πληροφορίες, αλλά πραγματικά εδώ έχουμε μπροστά μας αξιόπιστες πληροφορίες οι οποίες καταδεικνύουν ότι η ισότητα ε, των φύλων δεν είναι απλά μέρος αλλά αναπόσπαστο πραγματικά μέρος ε, της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι κάποια από τα στοιχεία που είναι πίσω από την πρωτοβουλία της ισορροπίας ιδιωτικής ζωής και εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτά που μας παρουσιάσατε. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε όταν βλέπουμε τις αντιδράσεις, όταν παρακολουθούμε τις συζητήσεις και την πρωτοβουλία για την ισορροπία ιδιωτικής ζωής και εργασίας, πολύ την υποστηρίζουμε και βλέπουμε ότι είναι καταστάσεις που είναι υποφελείς για όλους που είναι στο μέλλον και μας περιμένουν και έχουν φτάσει ήδη σε αυτή το πλαίσιο τα κράτη, κάποια κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι αντιδράσεις βλέπετε, συναντάτε όταν παρουσιάζετε αυτά τα στοιχεία στα διάφορα κροατήρια σαν πολιτικοί βρίσκουμε ακραίες θέσεις θετικές ή αρνητικές τίποτα στο μέσο των δύο αντιδράσεων. Και είναι αρκετά δύσκολες, είναι σκληρές οι συζητήσεις που γίνονται. Και έτσι αισθάνομαι, έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται χρόνος πριν δούμε διαφορά Υπάρχουν μία-δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στο σωστό δρόμο. Αλλά υπάρξουν τόσες χώρες που πρέπει να πολεμήσουν επί για να πετύχουν τους στόχους. Τι τους λέτε όταν τους συναντάτε αυτούς που έχουν αρνητική αντίδραση. Για την ισορροπία εργασίας και ιδιωτικής ζωής. διότι από αυτά που είπατε εκεί κατέληξα στο θέμα, στο πλαίσιο αυτός της της εργασίας με την ιδιωτική ζωή. Σε αυτό αναφέρεστε, με ένα διαφορετικό τρόπο. Τι ζητώ να μας, μας πείτε, υπάρχει ισχυρή αντίδραση, αρνητική. από τις διάφορες χώρες και τους θεσμούς, από τους λαμβάνοντες αποφάσεις. Πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση όταν υπάρχει μια τόσο έντονη αρνητική αντίδραση, είναι η ερώτηση. Απάντηση πρώτα απ' όλα, η ισορροπία εργασίας ιδιωτικής ζωής είναι σημαντικότατη η πρωτοβουλία και αρνητικές αντιδράσεις ίσως να δημιουργούνται από την ερμηνεία που δίνουν κάποιοι στο όλο μήνυμα και την προσπάθεια. Όταν αναλύσαμε τους διάφορους δείκτες, είδαμε ότι οι άντρες συνήθως εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες, κυρίως όταν έχουν οικογένειες με πολλά παιδιά. Και οι γυναίκες τους ή οι σύντροφοί τους δεν έχουν πολλές δυνατότητες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το να δουλεύει κανείς πολλές ώρες, πολύ σκληρά, για να βγάλει πολλά λεφτά, αλλά να μην είναι χαλαρή η ζωή του μετά οικογενειακή το βράδυ, να μην έχει τη δυνατότητα για ποιοτική ζωή με τα μέλη της οικογένειας, δεν είναι ένα θέμα που αφορά τη συμφιλίωση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, αλλά είναι κάτι που διαμορφώνει και την οτροπία οι άντρες χάνουν αν πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει και αυτοί να είναι μαζί με την οικογένειά τους. Ζουν λιγότερο. Μπορεί να έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας σε νεότερη ηλικία. Πολλά φαινόμενα συνδέονται με την αντίληψη της κοινωνίας και την οτροπία. Η ισορροπία εργασίας και ιδιωτικής ζωής είναι ένας βασικός παράγων που βοηθά να καλύψουμε τα κενά μεταξύ των φίλων σε συνάρτηση με πολλά άλλα στοιχεία. Προσωπικά πιστεύω ότι η πρωτοβουλία είναι καλή και θα μπορέσουμε όχι μόνο να δημιουργήσουμε πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, καλύτερη Ευρώπη, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και το δυναμικό το γυναικείο ε, που έχουν πολύ καλή παιδεία και αυξάνεται το επίπεδο παιδείας των γυναικών και μάλιστα σε σχέση με την παιδεία των ανδρών. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τη φιλοξενούμενή μας. Η κυρία Λίλιαν Μπικεβικιούτσε, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής μας των Γυναικών και καθυστέρησε. Ε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λυπάμαι πολύ για την καθυστέρηση. Δυστυχώς, κυρία Λάντμπακ, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την παρουσίασή σας. Θα έχουμε ε, την ευκαιρία να τα συζητήσουμε κατηδίαν αυτά τα θέματα για να μάθω περισσότερα για τη μελέτη σας. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ε, στα όσα είπε ο πρόεδρός μας για την πρωτοβουλία ε, για την ισορροπία μεταξύ εργασιακού και ιδιωτικού βίου. Είναι από τις βασικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το συζητάει το Κοινοβούλιο ε, αυτό για το πώς θα βελτιωθεί η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας πώς θα βρούμε τρόπους έτσι ώστε οι γυναίκες να επιστρέψουν στην αγορά ε, εργασίας για να μπορούν να έχουν δουλειά έτσι ώστε να εξασφαλίσουν και ψηλότερες συντάξεις μεθαύριο. Αυτό το συζητούν λοιπόν και τα κρατημέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα θέμα που απασχολεί. Στη Λιθουανία έχω συμμετάσχει σε πολλές συζητήσεις για αυτά τα θέματα και πολύ συχνά ακούω διάφορα επιχειρήματα ε, του τύπου ότι ε, πώς είναι δυνατόν να παίρνουν και οι άνδρες ε, γονική άδεια μέχρι τέσσερις μήνες, τι θα την κάνουν, πώς θα την αντιμετωπίσουν. Μερικοί το θεωρούν απαράδεκτο αυτό. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να αλλάξουν οι νοοτροπίες και οι ε, συμπεριφορές. Να ε, επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση, να αρχίσουμε από τον υπηαγωγείο, από το δημοτικό και να αλλάζουμε τις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες των ανθρώπων, να καταπολεμήσουμε τα παλιά στερεότυπα. Γιατί δεν αρκεί μια οδηγία, όσο καλή και να είναι. Δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση. Ούτε πρόκειται να επιφέρει ισότητα στις κοινωνίες μας. Η δε ισότητα στην αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Τι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε εμείς περισσότερο, πώς να επενδύσουμε καλύτερα ε, στην κοινωνία και στους πολίτες. Συμφωνώ πολύ με αυτό που λέτε. Πολλές φορές το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται με αλφαγιώτα μια οδηγία ή πώς ενθαρρύνουμε, πώς παροτρύνουμε τον κόσμο και όπως είπατε τα στερεότυπα, τα μοντέλα, τα, οι ρόλοι που αντιστοιχούν στον άνδρα και στη γυναίκα στην κοινωνία είναι ένα ζήτημα. Και πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες πιστεύουν ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει ο άνδρας ε, στο σπίτι, ας πούμε. Ακούμε διάφορα σχόλια ότι δεν μπορώ να αφήσω το μωρό μου μόνο του, ε, ε, το να θέσω στον άντρα μου. Δεν ξέρει να τα βγάλει πέρα, δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί. Και πολλές φορές ακούω ότι αυτή η γονική άδεια των τεσσάρων μηνών για τον πατέρα ε, είναι κάτι που δεν θέλουν οι οικογένειες. Γιατί συνήθως ο άνδρας αμείβεται περισσότερο και θεωρούν ότι είναι απώλεια εισοδήματος για την οικογένεια αυτή και δεν το προτιμούν. Εδώ πρόκειται για την οικογένειά μας. Εσύ αποφάσισες να κάνεις οικογένεια, εσύ ήθελες παιδιά είναι και το δικό σου μέλλον και δική σου ευθύνη αυτή, να αναλάβεις ευθύνη σου. Και έτσι αισθάνεσαι και καλύτερα. Ο τρόπος λοιπόν που μεταδίδουμε, που διαβιβάζουμε το μήνυμα έχει σημασία. Και καμιά φορά χρειάζεται να γίνουν συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης για να βοηθούν ιδιαίτερα του νέου άντρε να καταλάβουν ότι αυτοί θα χάσουν αν δεν πάρουν γονική άδεια. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, που ήρθατε. Είμαι ε, βεβαία ότι θα είμαστε σε επαφή μαζί σας για ερωτήσεις και απαντήσεις γιατί αυτό το θέμα ε, της ε, συμφιλίωσης του εργασιακού με τον ιδιωτικό βίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον και θέλουμε να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Λοιπόν, επόμενη συνεδρίαση 16 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας στις 3 το απόγευμα ε, με 3 με 6,5 και 19 Οκτωβρίου 9 το πρωί με Του των όλων λεχθέντων θα ήθελα να σας θυμίσω ότι έχουμε κοινή ακρόαση το απόγευμα με την Επιτροπή Πολιτισμού για το Ευρωπαϊκό ε, Σώμα Αλληλεγγύης. Είναι ένα θέμα σημαντικό και για τις δύο επιτροπές και για τη δική μας επιτροπή ακόμα περισσότερο. Να μην δημιουργήσουμε μια νέα παράλληλη αγορά εργασίας που δεν είναι αρκετά καλή για τους νέους μας. Καλό το σώμα αλληλεγγύης να δούμε περί τίνος πρόκειται και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα πώς θα οργανωθεί για να αποφυφθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αλλάζουμε κτίριο. Α1G3 στο κτίριο Σπινέλη θα αρχίσουμε στις 3 η ώρα. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι ε, στη συνεδρίαση αυτή. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Λέξη συνεδρίασης.